άλλαξε, εγκρίνεται. Προβλέπεται τώρα δήλωση του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποχώρηση του ΕΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω στου βουλευτέ ότι για τη συζήτηση αυτή δεν προβλέπεται διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ, ούτε θα γίνουν δεκτέ ερωτήσει βάσει τη γαλάζια κάρτα και του συστήματό τη. Πρώτη παρέμβαση. Η κυρία Τσιότ, εκ μέρους του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξότιμοι βουλευτέ, πριν από δύο εβδομάδε είδαμε τι ήδη έχει κάνει το Συμβουλίο κατόπιν τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη συμφωνία τη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κατόπιν τη εγκρίσεω τη πολιτική δήλωση. Εκεί όπου ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο για τις μέλουσες σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου του Νοεμβρίου. Αυτό έγινε αμέσω μετά αυτή τη τόσο σημαντική ψηφοφορία στο Westminster. Και πρόκειται για μια ψηφοφορία που είναι ατυχή, που μα λυπεί. Και ελπίζαμε ότι τουλάχιστον αυτό θα είναι ένα ξυπνητήρι, θα είναι σήμα κινδύνου, ούτω ώστε η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, το Ηνωμένο Βασιλείο, να συνέλθουν και να ξαναβρούν τη σωστή ρότα. Από ό,τι καταλάβαμε από τη ψηφορία όμως και τέτοιο δεν ισχύει. Και τώρα μάλλον η αβεβαιότητα έχει ενταθεί. Τι ρυθμίσεις εναλλακτικέ θα μπορούσαν να υπάρξουν όσον αφορά τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τη χώρα, πώς είναι δυνατόν αυτά να τα συγκεράσουμε. Ε, μια τέτοια ρύθμιση με μια ξεκάθαρη θέση δική μας ότι η συμφωνία της αποχώρησης είναι καλύτερος δυνατός συμβασμός. Αυτό το κείμενο το οποίο προέγγιψε από τις διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω τώρα να προβώ σε κάποιο είδου ε, ε, μαντεψιά για το τι θα γίνει σχετικά με αυτές τις προτάσεις, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, η άτακτη έξοδος γίνεται πιο πιθανή και οι συνέπειές της ε, θα καταστούν ακόμα χειρότερες για μας και ακόμα χειρότερες για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, οικονομική κύκλη όλο ένα και περισσότερο επισημαίνουν ε, αυτή την κατάσταση αβεβαιότητος και σε σχέση με την τροχιά πήραν τα πράγματα και σε σχέση με το τι γίνεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βρετανία και για τις θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν. Οπότε τώρα οδηγούμεθα σε περισσότερες ε, εντάσεις, συγκρούσεις και Όλα αυτά μας δοκιμάζουν όσον αφορά την ενότητά μας, την αποφασιστικότητά μας, γιατί θέλουμε να αντισταθούμε στον πειρασμό κάποιων διμερών ε, ρυθμίσεων. Για την άλλη μεριά υπάρχει ένας κοινό ε, στόχος όταν ε, τα αναγκαία κατεπιμένα μέτρα εγκριθούν η ευθύνη και η αρμοδιότητα είναι της κυβέρνησης της χώρας. Εμείς πάντως θέλουμε να βοηθήσουμε, θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της κύρωσης. Οπότε, σε σχέση με αυτό, μέσα στα όρια και στο πνεύμα των αρχών μας και των θέσεών μας, όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών και όσον αφορά το backstop, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε επαφές σε διευκρινήσεις, εάν αυτό βοηθάει τα πράγματα της διαδικασίας κύρωσης και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας δεν προβλέπεται. Επομένως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκαθαρίσει ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα κάνει και στο μεταξύ εμείς συνεχίζουμε την διαδικασία της ε, κύρωσης σε μας που ε, προχωράει παράλληλα με την διαδικασία που κουζδεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από, από πλευρά χρονικών ε, πλαισίων, πλευρά περιεχομένου, θα πρέπει να εισηγήσουμε την προπαρασκευή για κάθε δυνατό σενάριο, ακόμα και αν έχουμε έξοδο χωρί συμφωνία. Το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο, επομένω, έχουν εντείνει τι προσπάθειέ του, ε, τι προπαρασκευαστικές για καταστάσεις ε, έκτακτες ε, ούτως ώστε να υπάρχει ένα στέγανο πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ε, νέα νομοθεσία σε αυτή την ύστερη φάση από πλευράς νομοθετικών ερχών, αλλά πιστεύουμε ότι με την συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Και με ενθαρρύνει η συμφωνία που ήδη έχει κλείσει όσον αφορά τις προτάσεις σχετικές με το Brexit. Η Προεδρία, σε συνεργασία με εσά θα διευκολύνει το να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για κάτι που ανάγκη. γέρος. και σας ευχαριστώ πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Ρία. Επόμενος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής ο κύριος Ζωνκλόντι Γιούνκερ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε λιγότερο από 60 ημέρες το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια κακή απόφαση. Ακούστε, ακούστε. Ακόμα και ενώ η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπερασπιζόταν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα αυτό γινόταν με σεβασμό. Η συμφωνία αποχώρησης και η πολιτική ε, δήλωση που συμφώνησαν 27 και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το αποτέλεσμα. Η συμφωνία αποχώρησης παραμένει η μόνη και καλύτερη δυνατή συμφωνία. Αυτό το είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέμβριο, το είπε και το Δεκέμβριο, το είπε και τον Ιανουάριο, μετά από την πρώτη σημαντική ε, ψηφοφορία στη Βολή των Κοινοτήτων. Η συζήτηση και η ψηφοφορία εχθές στη Βολή των Κοινοτήτων δεν αλλάζουν το γεγονός αυτό. Η συμφωνία αποχώρησης δεν πρόκειται να τύχει επαναδιαπραγμάτευσης. Και οι δύο πλευρές έχουν διατρανώσει ότι δεν μπορεί να επανέλθει σκληρό σύνορο ε, στην ε, Ιρλανδία. Δεν πρόκειται να αλλησθήσουμε στους σκοτεινούς καιρούς του παρελθόντος. Πιστεύω την Πρωθυπουργό. Επίση, πιστεύω ότι χρειάζεται και ένα δίχτυ ασφαλείας που θα πρέπει να μας εξασφαλίζει απέναντι σε αυτό το κίνδυνο. Δεν έχουμε ούτε επιθυμία, ούτε ε, έναυσμα για να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο ασφαλείας. Αλλά κανένα δίκτυο ασφαλείας δεν θα είναι ασφαλές αν μπορεί να αφαιρείται ανα πάσα στιγμή. Καμιά φορά έχω την αίσθηση από καιρό σε καιρό ότι ορισμένοι ελπίζουν 26 ε, άλλες χώρες να εγκαταλείψουν το backstop και να αφήσουν μόνοι τους την Ιρλανδία την τελευταία στιγμή. Αλλά αυτό δεν είναι παιχνίδι, ούτε είναι διμερός απλώς το θέμα. Αγγίζει την ίδια την καρδιά το τι σημαίνει να είσαι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σύνορα της Ιρλανδίας είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων μας. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε από τη χθεσινή συζήτηση ότι η βολή των κοινοτήτων είναι κατά πολλών πραγμάτων είναι κατά του Brexit χωρίς συμφωνία, είναι κατά του Brexit έτσι κι αλλιώς, αλλά παρόλα αυτά δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς επιθυμεί η Βουλή των Κοινοτήτων. Υπέρ είναι. Η αρχή, ε, η έννοια των εναλλακτικών ρυθμίσεων δεν είναι καινούρια. Συζητήθηκε και στις διαπραγματεύσεις και αναφέρεται και στην πολιτική δήλωση και στην επιστολή μας προς την Πρωθυπουργό Μέη, ο πρόεδρος Τούσκ και ο υποφαινόμενος ε, δεσμευτήκαμε να το διερευνήσουμε περαιτέρω κατά προτεραιότητα. Αλλά η έννοια δεν είναι σχέδιο, δεν είναι επιχειρησιακή λύση. Πολλοί στη Βουλή των Κοινοτήτων και μεταξύ εκείνων που υπερψήφισαν και μεταξύ εκείνων που καταψήφισαν την τροπολογία ε, έχουν επίγνωση αυτού του γεγονότος. Εγώ θα εξακολουθήσω να είμαι σε στενή επικοινωνία και επαφή με την Πρωθυπουργό Μέη, την οποία σέβομαι και τιμώ απολύτως και θα ακούσω τις ιδέες της, αλλά θα είμαι και απολύτως ξεκάθαρος σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία σήμερα παρουσίασα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας πω ρητά ότι η χθεσινή ψηφοφορία ύφξησε τον κίνδυνο μιας άτακτης υποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια ε, συμπεριλαμβανομένου και του χειρότερου δυνατού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε την προετοιμασία της ε, το Δεκέμβριο του 2017 και τις τελευταίες εβδομάδες σε στενή συνεργασία με το Κοινοβουλίο σας κύριε Πρόεδρε επιταχύναμε τις προετοιμασίες μας. Έχω στείλει μια ομάδα σε κάθε πρωτεύουσα για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστήριξε την προσπάθεια αυτή από την αρχή ήδη. Αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, έχουμε κοινοποιήσει και δημοσιεύσει 88 κοινοποιήσεις για να δείξουμε τις ε, συνέπειες του Brexit σε διάφορα θέματα και 18 προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι τρεις τελευταίες αφορούν το πρόγραμμα Εράσμους, την κοινωνική ασφάλιση και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα εγκρίθηκαν και παρουσιάστηκαν. Θα ήθελα ήδη από τώρα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέχονται ε, έτσι ώστε να φτάσουμε σε σύντομα σε λύση για όλα τα επίγοντα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, περισσότερο από ποτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την ψυχραιμία της, την ενότητά της, την αποφασιστικότητά της, ε, όπως ε, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στην ε, υπόθεση αυτή υπάρχει ο εξή χρυσός κανόνας. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε την συμφωνία και την πολιτική δήλωση. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, εγώ είμαι εκφύσεως αισιόδοξο και παραμένω και πιστεύω στους δημοκρατικούς θεσμούς. Έτσι είμαι πεπισμένος και από πεποίθηση. Ε, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία και θα υπάρξει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί συγγνώμη, μου, με τη νέα μας ε, εταιρική σχέση. Νυχθημερών εργαζόμαστε για να ε, είμαστε έτοιμοι. Ό,τι και να γίνει, πάντα θα εξασφαλίσουμε ότι θα είστε οι πρώτοι ε, που θα μάθετε τι σημαίνει και οι τελευταίοι που θα αποφασίζετε. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον ε, επικεφαλής διαπραγματευτή κύριο Μισελ Μπαρνιέ, Θέλω να τονίσω και προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον επικεφαλής διαπραγματευτή για το Ευρωκοινοβούλιο, ποια και αν είναι η λύση του προβλήματος του Brexit, για μας η προάσπιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών 350.000 ε, που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι προτεραιότητα. Το ίδιο και για του Βρετανού πολίτε που κατοικούν σε εμά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ε, αυτή τη στιγμή λοιπόν μας ενδιαφέρουν το ίδιο οι Βρετανοί πολίτες όσο και οι δικοί μας που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Μπαρνιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, κυρία Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε ξανά εδώ στη Σύνοδο να παρουσιάσω εδώ τη θέσεις μου. Μέρα με τη μέρα μαζί με τον πρόεδρο Γιούνκερ προσπαθούμε να χτίσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, διαφάνεια στο διάλογο και την όλη συζήτηση που από κοινού οικοδομήσαμε μαζί σας, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, μαζί με τον κύριο Φερχόφστατ, μαζί με όλους τους συνεργάτες σε κάθε γύρο συζήτησης που έχουμε. Για πρώτη φορά η Πρωθυπουργό Τερέζα Μέη ζήτησε να ξανανοίξει η εξέταση της συμφωνίας αποχώρησης. Και εφόσον θα υπάρχει ψηφοφορία απόψε το βράδυ, υπάρχει και μια απόσταση πλέον σε σχέση με μια συμφωνία που ίδια είχε διαπραγματευτεί και επί της οποίας είχαμε καταλήξει σε συμφωνία. Η Βρετανική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την ανοιχτή της υποστήριξη στην τροπολογία του κυρίου Γκράμ Μπράντι, ο οποίος ζητά την αντικατάσταση του συστήματος backstop που είχαμε προβλέψει στο πρωτόκολλο για την Ιρλανδία με εναλλακτικές διευθετήσεις. Διευθετήσεις που σε καμία περίπτωση δεν έχουν αποσαφινιστεί ακόμη. Ταυτόχρονα η Βουλή των Κοινοτήτων απέρριψε το σενάριο της έλλειψης της απουσίας συμφωνίας, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να διευκρινιστούν οι τρόποι με τους οποίους θα αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο. Να, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα το απόγευμα. Στη διάρκεια αυτή της μακροσκελούς και ε, πέραν του συνηθισμένου ε, διαπραγμάτευσης. Και κύριε Πρόεδρε, όπως βρισκόμουν στις πρώτες γραμμές του αγώνα αυτού, ε, στο πλευρό του Προέδρου Γιούνκερ, Τούσκ και έσα του ιδίου, κάποια στιγμή θα πρέπει να πω ότι τα πράγματα ήταν και σοβαρά και δύσκολα. Χθε το βράδυ με τον κύριο Γιούνκερ ε, θυμήσαμε ότι συμμεριζόμαστε τη βούληση του Βρετανικού Κοινοβουλίου να αποφύγουμε την απουσία, την έλλειψη συμφωνίας και με την κυρία Μέη, ε, καλώς καταψηφίστηκε ε, το σενάριο του no deal. Αυτό όμως δεν το απαλήθηκε πλήρως το σενάριο αυτό. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, για μας η συμφωνία της αποχώρησης παραμένει και είναι το καλύτερο μέσο για να ε, προβλέψουμε μια τακτική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και με τρόπο έφτακτο να μπορέσει η να γίνει σεβαστή η τοποθέτηση τη πλειοψηφία των Βρετανών πολιτών να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί το σεβόμαστε. Πιστεύω ότι παρά τι σημερινέ δυσκολίε μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο υπό την προπόθεση ότι θα είμαστε ταυτόχρονα και ρεαλιστέ και διαυγεί στη σκέψη μα. Θα είμαστε πλήρη σεβασμού και θα αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Και η μεν και η δε. Μάλιστα, η μεν μαζί με του δε. Ε, ο μηχανισμός του backstop για τον οποίο μίλησε ο κύριος Γιούκερ είναι μέρος της συμφωνίας αποχώρησης και η συμφωνία αυτή δεν μπορεί να ξαναγίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου που ε, συμπίπτουν πλήρως με τις δηλώσεις και τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου για το θέμα δεν αφήνουν να ε, υπάρξουν εδώ αμφιβολίες. Θέλω να πω δύο κουβέντες για το μηχανισμό backstop ώστε όλοι να αντιληφθούν πλήρως περί τίνος πρόκειται. Ο μηχανισμός backstop δεν είναι δογματική απόφαση, είναι μια λύση, μια ρεαλιστική λύση που προσφέρεται. Επιζητήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και υπό τον πλήρη ελεγχό σα να εξεύρουμε λύσεις σε προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όλος ιδιαιτέρως, αλλά όχι μόνον, στη Βόρεια Ιρλανδία με την προοπτική του Brexit ο μηχανισμός backstop, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία Αποχώρησης, είναι το αποτέλεσμα, το πόρισμα αυτών των ε, εντατικότατων διετών ε, διπλωματεύσεων που έχουμε ε, διενεργήσει μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και ποτέ κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μια ρεαλιστική απόκριση για το τι θα γίνει με την ίσο της Ιρλανδίας εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε με την πλήρη του εθνική κυριαρχία να αποχωρήσει όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Ενιαία Αγορά και την Τελωνιακή Ένωση χρειάστηκαν δύο χρόνια για να βρούμε αυτή τη λύση. Λύση που ε, επιτρέπει να συγκεντρωθούν και να ικανοποιηθούν πολλές προϋποθέσεις ταυτόχρονα. Πρώτη, να αποφύγουμε την, ε, ε, το νέο σκληρό σύνορο μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλαδή να σεβαστούμε τις συνθήκες ειρήνης, διαλόγου και συμφιλίωσης που επικρατούν εδώ και 20 χρόνια στην ίσο της Ιρλανδίας. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής στο Belfast θυμίζω ότι το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο με την ε, ψήφο της Πρωθυπουργού του επανειλημμένος επανέλαβε την δέσμευσή του να παραμείνει συνεγγύητη της ε, πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας αυτής της Μεγάλης Παρασκευής και με το πρόγραμμα PIS, με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, με τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές, με τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό εδώ και χρόνια, φροντίζουμε να είναι ε, ομαλή η συνεργασία και η συνύπαρξη των διαφορετικών κοινοτήτων στην Ιρλανδία. Πρώτη προπόθεση αυτή. Δεύτερη, η βούληση, το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου, τη κυβέρνησή του, να παραμείνει η Ιρλανδία, ε, η Βόρειο Ιρλανδία, ένα ξεχωριστό, ε, μια ξεχωριστή επικράτεια του κράτου. Τρίτη προπόθεση, κάτι που ε, για το οποίο είμαστε όλοι συλλογικά υπεύθυνοι διασφάλιση και η προφύλαξη τη ε, ενιαίας αγορά. Αυτό για μα, κύριε και κύριοι είναι καθοριστική σημασία. Τα ευρωπαϊκά σύνορα, επειδή το θέλησε το Ηνωμένο Βασίλειο, θα γίνουν σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί θα σταματούν τα σύνορα τη εσωτερική αγορά. Θα είναι τα νέα μα εξωτερικά σύνορα. Άρα, αυτό που διακυβεύεται είναι η προστασία όλων των καταναλωτών και όλων των επιχειρήσεων της Ένωσης. Για να το πω πολύ πιο σταράτα, η απόφαση του ΕΒ Βασιλείου να φύγει από, το Βασι... από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ένωση της Εσωτερικής Αγοράς έχει και πρακτικές συνέπειες το κάθε εμπόρευμα, το κάθε αγαθό, το κάθε ε, ζωντανό ζώο, το κάθε προϊόν ζωική ή φυτική προέλευση που έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινώντα από το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι απλώ περνάει στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ιρλανδία, αλλά μπαίνει στην εσωτερική αγορά, στην εσωτερική αγορά των δικών σα των χωρών φύση, η ποιότητα, η ασφάλεια και η νομιμότητα των προϊόντων αυτών. Η ασφάλεια για την ε, προστασία των ζώων και το λέω γιατί αφορά του υπουργού γεωργία και κτηνοτροφίας των χωρών μα. Όλα αυτά απαιτούν ελέγχου. Ελέγχου που κάνουμε σε κάθε σημείο των εξωτερικών μα σύνορων παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελέγχους τελωνιακούς, υγειονομικούς, οικονομικούς, κτηνιατρικούς και νομικούς Αυτήν την προστασία την οφείλουμε σε όλους μας τους καταναλωτές. Τα 507 εκατομμύρια μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, τα 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις μας. Το οφείλουμε σε όσους ζουν και εργάζονται στην εσωτερική αγορά. Ιδού. Και μεταξύ όσων σήμερα ζητούν την ε, αναστολή, την απάλληψη του μηχανισμού backstop, υπάρχουν και Βρετανοί βουλευτέ. Μίλησα σήμερα, με, σήμερα το πρωί με έναν από αυτού. Είναι σημαντικό να διαπραγματευτούν μαζί μα γνωρίζουν ότι ο μηχανισμός backstop όμως είναι η λύση που καταφέραμε με δυσκολία να βρούμε γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ είναι η, ε, ε, η προστασία της καρδιάς της Ευρώπης βρίσκεται στην καρδιά των υποχρεώσεων και των αρχών μας, δηλαδή την προστασία της εσωτερικής αγοράς σε όλες τις, τις διαστάσεις και τις προεκτάσεις. Δίκαιο για τις εταιρείε και δικαιώματα των καταναλωτών, για τις επιχειρήσεις, για το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας. Για να είμαι ειλικρινή, όταν ακούω κάποιου που συμμετείχαν και όλα τι διαπραγματεύσει να εκφράζονται όπω τοποθετήθηκαν, ε, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να δεχτώ αυτό το εγκεφαλικό παιχνίδι και τη χειραγώγηση που προσπαθούν να παίξουν. Το παιχνίδι κατηγοριών που προσπαθούν να παίξουν. Και εδώ δεν είναι τόσο απλό ε, να πούμε ότι θα αφήσουμε στην τύχη του το, την εσωτερική αγορά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να κινδυνεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε και εναλλακτικέ διαθετήσεις, όπως αυτές που αναφέρθηκαν χθε από την Βουλή των Κοινοτήτων Ακούσαμε και τη Βουλή τη Ιρλανδία και τι πολιτικέ δηλώσει. Και τα είπε και ο πρόεδρο Γιούγκερ. Θα είναι προτεραιότητα στι μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε εντατικά αμέσω μετά την υπογραφή τη Συμφωνία Αποχώρηση. Σήμερα όμω, κανεί ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη δεν είναι σε θέση να προβλέψει ε, ξεκάθαρα και κατά ποια θα είναι η φύση αυτών των εναλλακτικών διευθετήσεων. Εάν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Εάν θα ε, πλέον ε, ε, απόλυτα του ίδιου στόχου με το μηχανισμό backstop. Αυτά θέλω να σα πω. πλήρη διαυγεία και ε, ηρεμία. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αυτό είναι το σχέδιο συμφωνία που σα προτείνουμε να κυρώσετε και χρειαζόμαστε το μηχανισμό backstop ω έχει. Εάν απορριφθεί στη σημερινή του μορφή, ουσιαστικά απορρίπτεται η λύση που έχουμε εξεύρει μαζί με τους Βρετανούς. Και το πρόβλημα θα παραμένει όπως το περιέγραψα. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα και πέραν των εναλλακτικών διευθετήσεων που επίσης υπενήθηκα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπως και το Ευρωκοινοβούλιο ήδη επανειλημμένος και σαφώς απέρριψαν την ιδέα να υπάρξει χρονική, ε, χρονικό όριο ή μονομερής απάλληψη του μηχανισμού backstop διότι σε αυτή την περίπτωση θα αλλοιωνόταν απευθείας η ίδια η φύση του backstop. Δεν θέλουμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε ε, είναι ένα μηχανισμό ασφαλεία που υπάρχει γιατί πρέπει να υπάρξει. Όπω και εσεί έχετε ασφάλεια για τα σπίτια σα, τα διαμερίσματά σα, είναι κάτι που χρησιμοποιείται εφόσον χρειαστεί. Η συμφωνία λοιπόν αποχώρηση, την οποία συζητούμε και την οποία πολύ καλά γνωρίζετε, πάει πολύ μακρύτερα από το θέμα τη Ιρλανδία. Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει τα δικαιώματα 4,5 εκατομμυρίων πολιτών. Κύριε Ταγιάννη, αναφέρατε την προτεραιότητα του Κοινοβουλίου. Είναι και δική μα από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Και ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν γίνει η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ε, συμπολιτών μα, των συμπατριωτών μα, 3,5 εκατομμυρίων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τι διαφορετικέ μα χώρε είναι ε, προτεραιότητα. Το ίδιο και για το 1,5 εκατομμύριο Βρετανών που ζουν στι χώρε μα. Παραμένει προτεραιότητα η διασφάλιση των δικαιωμάτων του. Επίση, προστατεύουμε το σύνολο των δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού και στι 28 χώρε μέλη. Οι δεσμεύσει που αναλάβαμε όταν ήμασταν 28 θα πρέπει να γίνουν σεβαστέ και μετά. Ε, το ίδιο και για τη μετάβαση του, ε, της διάρκειας 21 μηνών για τις επιχειρήσεις και τις ε, διοικητικές υπηρεσίες. Ώστε και από τις δύο πλευρές να ε, είμαστε προετοιμασμένοι και οι μελλοντικέ σχέσει να μπορούν να εξομαλυνθούν. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να διαπραγματευτούμε και αυτέ τι μελλοντικέ σχέσει. Πρέπει να περάσουμε από νέε φάσει, νέα κύματα διαπραγματεύσεων. Αυτή η συμφωνία λοιπόν είναι μια προπόθεση για να δημιουργηθεί και να οικοδομηθεί το κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ μόν και του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια χώρα που θα παραμείνει φίλη, σύμμαχο, εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μια πραγματική εταιρική σχέση, ε, ακλόνητη και σταθερή. Για τις μελλοντικέ αυτές σχέσεις, οι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι και θα παραμείνουν πρόθυμοι τις ερχόμενες ημέρες να δείξουν ακόμη μεγαλύτερη φιλοδοξία, να εργαστούν επί της ποιότητας και της, εντατικό, της έντασης που θα έχουν οι μελλοντικέ μας ιδίως οικονομικές σχέσεις. Και το γνωρίζετε κυρίες και κύριοι βουλευτές. Υπάρχουν πολλά μοντέλα συνεργασία που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Μοντέλα οικονομική συνεργασία με άλλε χώρε, τρίτε χώρε. Το καθένα από αυτά τα μοντέλα πρότυπα έχει διαφορετική εξισορρόπηση δικαιωμάτων υποχρεώσεων, αλλά υπάρχουν πολλά. Και απλώ να πω ότι αν τα βρετανικά αιτήματα εξελιχθούν και ξεπεράσουν το θέμα της, ε, την περίπτωση της απλής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, είμαστε και θα είμαστε προθυμότατοι να συζητήσουμε το οποιοδήποτε από αυτά τα μοντέλα για να δούμε τι νέε φιλοδοξίε μπορεί να εκφράσει η βρετανική πλευρά που θα ανταποκρίνεται και στι δικέ μα τι φιλοδοξίε. Όπω είπατε και εσεί και όπω έχουμε πει και εμεί και θα πει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι με πλήρη διάβια και ρεαλισμό, κυρίε και κύριοι, όπω κάνατε και εσεί, κυρία Υπουργέ, Βρισκόμαστε λιγότερο από 60 μέρε από την τελική προθεσμία, τη λήξη τη προθεσμία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, μέχρι τώρα ήταν η στάση τη Βουλή των Κοινοτήτων θετική για την λύση που ε, είχε προταθεί και ήταν παραδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπε και ο πρόεδρο Γιούγκερ λοιπόν, είναι ε, επίγον και αναγκαίο να προετοιμαστούμε για όλα τα δυνατά σενάρια και να προβλέψουμε όλα τα έκτακτα μέτρα, τα contingency μέτρα που μπορεί να χρειαστούν για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπω διαμορφώνεται μέσα από τη δική μα συνεργασία. εργασία, την εργασία των Πρόεδρων, των συνεργατών σα και όλου του ε, συνεργάτε μα στα κράτη-μέλη. Σα ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη σα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαριέ. Ε, μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτο, ο κύριο Μπροκ, εκ μέρου του ΕΛΚ. Herr Präsident, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύρια Προεδρεύουσα, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητέ Μισελ Μπανιέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχά τον Ζαν Κλοντ Ιούνκερ και τον Μισελ Μπαρνιέ για την καλή συνεργασία, την πραγματική διαφάνεια, την ενημέρωση που είχαμε, αλλά και το γεγονό ότι μα άκουγαν. Καλό παράδειγμα αγαστή συνεργασία. Και εδώ ερχόμαστε να το συνειδητοποιήσουμε πάρα πολύ καλά ότι στηρίζουμε αυτή τη διαπραγματευτική στρατηγική. Εχθές ζήσαμε μια ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων όπου απέρριψαν κάθε ε, λογική λύση για το νέο δημοψήφισμα, για την Τελωνιακή Ένωση. Το μόνο που συμφωνούν είναι να στείλουν ε, στις Βρυξέλλες για τρίτη τέταρτη φορά την κυρία Μέη να μιλήσει για το backstop, ουδέν νεότερον. Είναι πολύ σημαντικό τώρα πριν έρθει εδώ η κυρία Μέη επιτέλους να μιλήσουν μεταξύ τους. Είναι σκάνδαλο να μην μιλάει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης με την Πρωθυπουργού τρία χρόνια και παραπάνω. Όταν θες να βγεις πρέπει να ξέρεις ε, τι σε περιμένει πριν επιβαρύνεις τους άλλους. Ελάτε με μία ενιαία θέση, μιλήστε μεταξύ σας, φέρτε μια επικοδομητική ιδέα και λύση στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς είμαστε ενωμένοι, εσείς δεν είστε ενωμένοι. Κυβέρνηση, τόριδες, Labour είναι διχασμένοι. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ. Έχουμε αρνητική πλειοψηφία που απαρτίζεται από διάφορες ομάδες. Από τους σκληροπυρηνικούς του Brexit μέχρι εκείνους που είναι υπέρ της παραμονής και αυτοί μπορούμε να προτείνουμε οτιδήποτε, δεν θα ψηφίσουν αυτοί που θέλουν το Brexit, είναι σκληρό, και εκείνοι που ελπίζουν να παραμείνουν. Ορισμένοι θα απορρίπτουν τα πάντα όσο δεν είναι δημοψήφισμα. Αυτούς τους καταλαβαίνει η καρδιά μου, αλλά το μυαλό μου όχι. Και η κυρία Μέι να διαπραγματευτεί ένα οποιοδήποτε backstop, το ίδιο θα το απορρίψουν για τους ε, γνωστού λόγους. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η Ιρλανδία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε μεγάλη συμμετοχή στη συμφωνία ε, της Μεγάλης Παρασκευής. Θυμάμαι το φίλο μας και παλιό συνάδελφο, τον Τζον Χιούμ, που από εδώ από το Κοινοβούλιο κατέβαλε κάθε προσπάθεια να το κάνει. Και εμείς θα το υπερασπιστούμε και το πρόγραμμα για την ειρήνη. Δεν θέλουμε σκληρά σύνορα εκεί. Αλλά Όπω είπε και η Βρετανική κυβέρνηση, υποτίθεται δεν θέλει και αυτή η σκληρά σύνορα και επανειλημμένα υπέγραψε ότι θέλει backstop το Δεκέμβρη του 2017 για πρώτη φορά. Αυτά πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα. Εμείς θα υπερασπιστούμε την Ιρλανδία και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα μαλακό σύνορο. Αλλά θα πρέπει να έχει και την προθυμία του άλλου. Και το σημερινό backstop με αυτή την τελωνιακή ένωση είναι μια βρετανική εφεύρεση, βρετανική πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάνει άλλε προτάσει. Δηλαδή θέλουν να διαπραγματευτούν κάτι το οποίο πρότειναν οι ίδιοι. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί. Μιλήστε μεταξύ σας. Στο Λονδίνο και λύστε το μεταξύ σας. Και αν έχουμε την ε, συμφωνία αποχώρησης, υπάρχει και μεταφατική ρύθμιση, όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε πάρα πολλά πράγματα που εκκρεμούν. Νορβηγία, Ελβετία, ό,τι θέλετε συζητάμε για τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά γι' αυτό δεν χρειάζεται backstop. Κατά 99% στη μεταβατική περίοδο ε, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το backstop δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα στην ουσία. Αυτοί δεν θέλουν συμφωνία για τους διάφορους λόγους δικούς τους που σας ανέφερα. Λοιπόν, θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Βεβαίως, ε, τώρα είμαστε προετοιμασμένοι με την νομοθεσία και είναι σημαντικό ότι είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε αν έρθει πρόταση για να βρεθεί λύση. Θα καλωσορίζω όλα αυτά. Αυτό που είπε η Βολή των Κοινοτήτων, το ότι δεν θέλουν σκληρό Brexit, ούτε εμεί το θέλουμε. Καλά, εγώ δεν θέλω να φύγουν έτσι κι αλλιώ. Έτσι για να ξεκαθαρίσω τα χαρτιά μου και να τα ανοίξω. Αλλά είναι βρετανική απόφαση. Τι να κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε Και να περιορίσουμε όσο γίνεται τι ζημίε εκατέρωθεν. Αλλά για μένα είναι ξεκάθαρο, θα πρέπει να το γνωρίζει και ο λαό τη Βρετανία. Η ζημιά για το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πάντα μεγαλύτερη. Η ευρωπαϊκή ε, αγορά είναι 16 φορέ μεγαλύτερη από το Ηνωμένο Βασιλείο. Και όσοι παράγουν για την ευρωπαϊκή αγορά θα σηκωθούν να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα είναι μια πικρή ώρα αυτή που θα ζήσει η Βρετανία. Ελάτε να τα βρούμε, ελάτε να συμφωνήσουμε, αλλά θα πρέπει η Βρετανική πλευρά να έχει μία θέση και επικοδομητική. Ευχαριστώ πολύ. Excellent German from the British bench there. Thank you. Εξαιρετικά τα γερμανικά της, της ε, βρετανικής πλευράς εκεί. Επόμενος ομιλητής εδώ, κύριος Γκουαλτιέρη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητέ Μισελ, είναι δύσκολο να πει κανείς ότι δεν βρίσκεστε με μιας περίπλοκη δύσκολη καταστάσεως και ότι δεν έχει αυξηθεί ο κίνδυνος του νόντιλ. Η Βουλή των ε, Κοινοτήτων ε, ψήφισε. Δεν θέλει το ένα νόντιλ. Αυτό είναι καλό. Ταυτόχρονα όμως ζήτησε το backstop να αντικατασταθεί με εναλλακτικέ ρυθμίσεις το οποίο δεν προβλέπεται και είδαμε επίσης η ίδια από την που πριν από λίγες εβδομάδες μας είπε ότι το καλύτερο backstop ήταν ένα απόστασμα τμήμα της ε, καλύτερης δυνατή συμφωνίας τώρα, τώρα ζητεί την αντικατάσταση αυτού αυτό ε, έχει φέρει ε, συμπαράταξη και απέφυγε το διχασμό στο κόμμα της, αλλά έχει μπλοκάρει την κατάσταση. Θα πρέπει να ξαναεξηγηθεί εκείνη γιατί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στην εντολή τους προς το διπραγματευτή ξεκαθάρισαν ότι ένα λειτουργικό και δεσμευτικό backstop είναι στο τμήμα της συμφωνίας. Οπότε δεν θα δώσουμε το πράσινο φως σε κανένα deal χωρίς ε, τον backstop να μπορέσουμε να μην έχουμε κλειστά στην Ιρλανδία, να συνεχιστεί η ειρήνευση εκεί, η ειρήνη εκεί να διασωθεί. Αυτό δεν είναι μικροπολιτική και οπότε αυτό είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Και το backstop αποτελεί μια εγγύηση, αποτελεί μια επιλογή, μια τελευταία λύση και είναι αναγκαίο για να εξασφαλίσουμε ότι εάν έχουμε μια συμφωνία για τι μέλου μα με τον Βασιλείο δεν υπάρξει μέχρι το τέλο τη περίοδου, τότε τα ελάχιστα διασφαλιστικά μέτρα θα πρέπει να ισχύσουν για να μείνουν ανοιχτά τα σύνορα και έτσι να διασωθεί η αγορά. Και δεν χρειάζεται να σα επαναλάβω ότι έχει αλλάξει τον το πετήσει των Βρετανών και αυτό δεν ήταν μια εύκολη παραχώρηση από πλευρά μα. Το κάναμε όμω για να επιτρέψουμε στην Βόρεια Ιρλανδία να μείνει τμήμα τη ίδια τελειωνική επικράτεια όπω το υπόλοιπο Βασίλειο και έτσι να μην έχουμε ποσοστώσεις, ε, ελέγχους, δασμούς και αυτό το, το, το, το συμφωνήσαμε παρά το ότι είχαμε την αρχική πρόταση η οποία ήταν δίκαιη, απλή και δεν, δεν επέβαλε κάποιο είδους ε, περιορισμούς ε, στο εμπόριο της θάλασσας της Ιρλανδίας. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να υπάρχει ένα τέτοιο νοντήλ. Φυσικά το Νότιλ είναι κακό για όλες τις πλευρές, αυτό θα ήταν ένα ναυάγιο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ορθώς οι ευρωβουλευτές ξεκαθάρισαν, συγγνώμη οι βουλευτές είπαν ε, ότι αυτό δεν το δέχονται και επαναλαμβάνουμε σήμερα για άλλη μια φορά ότι θέλουμε να υπάρξει όσο γίνεται πιο στενή σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. πρόκειται για κόκκινη γραμμή του Ηνωμένου Βασιλείου που μέχρι τώρα μας ε, εμπόδιζε. Αυτό για μας σημαίνει ότι η μόνη εναλλακτική στο backstop είναι μια στενότερη σχέση με την χώρα. Οπότε αν θέλετε να εξασφαλίσουμε το να μην επικαλυστεί κανείς το backstop, τότε φτιάξτε μια θετική πλειοψηφία για μια πιο φιλόδοξη σχέση για τελωνιακή ένωση και κάποιο είδου καλύτερη ευθυγράμμιση με την ενιαία αγορά. Λιγότεροι από δύο μήνε απομένουν ε, μέχρι την αποχώρηση. Κατεπηγόντω θα πρέπει να δούμε μια επικοδομητική πρόταση από το Ηνωμένο Βασίλειο για να σταματήσει η εμπλοκή. Αλλιώ θα πρέπει να ξαναρωτηθεί ο Βρετανικό λαό αν χρειαζόνται περισσότερο χρόνο και σε αυτό είμαστε νυχτοί. Αλλά χρειάζεται ένα ξεκάθαρο πλάνο, μια ξεκάθαρη πρόταση για το πώ αυτό θα βοηθήσει. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε μια παράταση για ψεύτικες ε, υποσχέσεις ε, και τα λοιπά. Εμείς είμαστε ε, συνασπισμένοι, είμαστε συσπηρωμένοι. μπροστά έχουμε τον διαπραγματευτή μας, ξεκάθαρη εντολή και θα ακούσουμε τι θα πει και ό,τι έχει πει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενότητα. Ανησυχούμε, αλλά και είμαστε αισιόδοξοι ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ, Φόξ, για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστάς. Παρακαλώ να σέβεσαι τους ομιλητές, κύριε Κόμπεν. Κύριε Φόξ, ελπίζω και να σας δείξουν τον ίδιο σεβασμό. Κυρία Πρόεδρε, άκουσα πέντε ομιλίε ω τώρα σήμερα το απόγευμα που περιγράφουν τι προσπάθειε διαπραγμάτευση για τη Συμφωνία Αποχώρηση και πόσο καλή είναι. Όμως είμαι βέβαιος ότι θα έχετε προσέξει όλοι ότι αυτή η ίδια συμφωνία αποχώρησης απερίφθη πριν από δύο εβδομάδες στη Βουλή των Κοινοτήτων με συντριπτική πλειοψηφία. Γι' αυτό τώρα δεν είναι στιγμή να ευχαριστούμε τους αυτούς μας με, με ρητορικά σχήματα, αλλά πρέπει να συλλογιστούμε σοβαρά. Ήταν δύσκολο να απεμπλακεί το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως τώρα ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας είναι ξεκάθαρος, εφόσον επιλέξουμε να τον ακολουθήσουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν εδώ κάποιοι, όπως ο κύριος Μπροκ, που ελπίζει, ακόμα ελπίζουν ότι το Εμένο Βασίλειο θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζουν θέσει που εκφράζουν αυτή την ελπίδα. Όμω αυτό δεν είναι γραφτό να συμβεί. Είναι απλώς, ε, θα ήταν μάλλον απλώ ε, εξωφρενικό και παράλογο να αγνοήσουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο. Και δεν υπάρχει πλειοψηφία στην Βουλή των Κοινοτήτων υπέρ μια τέτοια επιλογή. Η πρόταση για να διοργανωθεί δεύτερο δημοψήφισμα απεσύρθηκε διότι ε, τύχανε τόσο λίγη υποστήριξη. Η Βρετανική κυβέρνηση και η Βουλή των Κοινοτήτων θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο έφτακτον και με συμφωνία. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε τα του πρωτοκόλλου της ε, Βορείου Ιρλανδίας Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να υποστηρίξουμε τη συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή. Όμω είναι παράδοξο το γεγονό ότι ο μηχανισμό του backstop που σκοπό έχει να αποφύγει το σκληρό σύνορο, ίσω μέσα σε 58 μέρε να γίνει το αίτιο δημιουργία ενό τέτοιου σκληρού σύνορου στην ίσο τη Ιρλανδία. Να επαναλάβω, ο μηχανισμός backstop στην τωρινή του μορφή δεν θα αποφύγει τη δημιουργία σκληρού συνόρου ίσα ίσα θα το δημιουργήσει. Γι' αυτό λοιπόν ας σταθούμε όλοι δύο λεπτά και ας συλλογιστούμε. Ίσως να είναι εύκολο να καθόμαστε σήμερα και να προασπιζόμαστε χειροκροτώντας την άκαμπτη προάσπιση μιας ήδη καταγεγραμμένης θέσης. Η ιστορία όμως δεν θα είναι τόσο ευγενική μαζί μας, διότι όπως έχουν τα πράγματα συμφωνία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συμφωνία εκτός και οι δύο πλευρές την έχουν εγκρίνει βάσει του νόμου τους. Οπότε δεν αρκεί να επαναλαμβάνουμε μέχρι αηδία ότι η συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Αυτό θα οδηγήσει σε συμφωνία μηδέν. Και όπω επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα οδηγήσει και σε σκληρό σύνορο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδία. Οπότε ελπίζω ότι ακόμη και σε αυτή την τελευταία στιγμή προσθήκες και αλλαγέ μπορούν να γίνουν ώστε να πάρουμε επιτέλους μια καλή συμφωνία και να την πάμε στην Βρετανία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, όπως είπε και ο κ. Μπαρνιέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει έναν εναλλακτικό τρόπο για να διεξαγάγει ελέγχους και εποπτεία χωρίς να υπάρχει νέο σύνορο. Να το δούμε τώρα λοιπόν αυτή την αυτή την, τον εναλλακτικό τρόπο. Α σκεφτούμε τι μηχανισμού και τι χρονικά όρια μπορούμε να βρούμε ω λύση. Α προχωρήσουμε με καλή προαίρεση. Έχουμε δείξει διαλλακτικότητα και γενναιοδορία. Α μην υποχωρήσουμε και φανούμε αδύναμοι, αλλά α φανούμε δυνατοί. Αυτό που αυτή τη στιγμή διακυβεύεται δεν είναι απλώ το σχέδιο συμφωνία, είναι η μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου ας βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια μελλοντική σχέση που θα επιτρέπει να καλλιεργούμε τις κοινέ μας αξίες, τα κοινά μας συμφέροντα και αυτό σε ένα κόσμο βεβαιότητας. Ας βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα για τους ε, φιλελεύθερους και δημοκράτες ο κ. Φερχόφστατ. Μετά τη χθεσινή ψηφοφορία η κυρία Μέη ανακοίνωσε ότι θα έρθει στις Βρυξέλλες και να σας πω ειλικρινά την ε, δική μου την ε, θέση, είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Ας έρθει και στο Ευρωκοινοβούλιο επιτέλους. Το έχουμε ζητήσει επανειλημμένος πριν από περισσότερο από ένα χρόνο. Το ερώτημα όμως είναι γιατί έρχεται, τι σκοπό έχει, τι θα κάνει θέλει να αλλάξει τις κόκκινες γραμμές, τις απαγορευτικές γραμμές της Βρετανικής κυβέρνησης, τις οποίες έχει παραμείνει η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα. Θα αλλάξει η έκβαση της, της διαπραγμάτευσης, της όλης διαδικασίας. Και η δεύτερη ερώτησή μου, η δεύτερη παρατηρήσή μου είναι τι εντολή θα έχει. Διότι προς στιγμή πρέπει να σας πω κύριε Φόξ ότι έχω ή τουλάχιστον μέχρι χθε δεν είχα δει το κοινοβούλιο σας να δίνει μια σαφή εντολή στην Τερέζα Μέη. Ψηφίσανε κατά ε, μια σειρά πραγμάτων κατά της συμφωνίας, κατά της μηδενικής συμφωνίας, κατά του backstop, όμως ως σήμερα έχουν περάσει δύο χρόνια και η Βουλή των Κοινοτήτων δεν έχει ψηφίσει ούτε μία πρόταση υπέρ κάποιου πράγματος υπέρ του ενό ή του άλλου, υπέρ πέρμια σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ. Τους τελευταίους δύο μήνες πρέπει να σας πω ότι πραγματικά εξαντληθήκαμε. Εξαντληθήκαμε. Όχι μόνο από την άλλη πλευρά της μάχης, και εδώ. Ατελείωτες συζητήσει. μακροσκελέστατη κατάλογη τροπολογιών, τροπολογίε που πήγαιναν δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, που τι επέλεγε ο πρόεδρο και χαθήκαμε για μια ελάχιστη διαφορά στην πλειοψηφία. Να σας να φέρω κατάλογο. 4 Δεκεμβρίου τροπολογία Γκριφ, η οποία ήταν ε, υπέρ του Remain. 22 η τροπολογία Google, η οποία πέρασε στις 8 Ιανουαρίου, ε, χάθηκε για 7 ψήφους. Μετά μια άλλη ε, τροπολογία, με 23 ψήφους χάθηκε, η τροπολογία Brady, η τροπολογία υπέρ του Live. Μία προς 16 χθε ε, και ε, μια πάλι μια τροπολογία Remain, η Spellman, ε, η οποία ήταν να μην υπάρξει καμία συμφωνία επιτάπητος. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα, έτσι θα λυθεί το πρόβλημα αυτών των διαστάσεων. Με αυτή τη συμπεριφορά, με αυτή τη διαδικασία, κάθε μέρα μεταβάλλετε τη στάση σας και τις απόψεις σας και δημιουργείται ένα κλίμα αβεβαιότητας, ανασφάλειας, αντί να οδηγείται σε, κάποιο, ε, σε κάποια τελική έκβαση η μελλοντική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματικά βλέπω τι συμβαίνει και δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω κάτι που ξεκίνησε σαν ένας τσακωμός και μαλλιοτράβηγμα στο κόμμα των συντηρητικών έχει γίνει υπαρξιακό πρόβλημα για όλη τη Βρετανία. Η τροπολογία Σπέλμαν χθε καταψηφίστηκε με 8 ψήφου, που έλεγε, μάλλον πέρασε η τροπολογία Σπέλμαν που έλεγε ότι είναι, αποκλείεται να μην υπάρξει καμία συμφωνία. Και αποσύρει την πρόταση αυτή και ήρθε πέντε λεπτά μετά η Πρωθυπουργό και είπε ότι όχι, αυτό δεν αποκλείεται. Είναι ένα σενάριο που μπορεί να συμβεί το μηδενική, η μηδενική συμφωνία. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Υπάρχει απουσία βεβαιότητα, απουσία διάβγεια. Και αυτή τη στιγμή, καθώ μιλάμε, λαμβάνει η χώρα μια συνάντηση μεταξύ του κ. Κόρμπιν, του επικεφαλή αντιπολίτευση και τη Πρωθυπουργού κ. Μέη. Ελπίζω κάτι να αποφασίσουν κάτι να συζητήσουν που να έχει περιεχόμενο. Όχι μόνο να τρώνε μπισκέ, μπισκότα ε, βουτώντας τα στο τσάι του το απόγευμα. Διότι θα θέλαμε μια λύση στο πρόβλημα. Θα ήταν λύση αν άρχιζαν να συνεργάζονται για μια διακομματική προσέγγιση. Μπα και μάθουμε κι εμεί ποια είναι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στο μέλλον. Δεν την γνωρίζουμε ακόμα. Κύριε Φόξ, θα πρέπει πρώτα να μπει η χώρα σας και μετά τα κόμματα. Πρέπει να μας πείτε ως χώρα πώς βλέπετε τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασίλειου. Όχι να χρησιμοποιείτε και να κάνετε κατάχρηση της ύπαρξης του Brexit για να ε, προχωράτε σε διελκυστήμβες δύναμες μεταξύ εσάς των ιδίων. Και η Πρωθυπουργός Μέη ας έρθει, να έρθει στις Βρυξέλλες ε, να μας πει ποια είναι η πλειοψηφία του κόμματό τη και τι θέλει για τη μελλοντική μα σχέση αυτή η πλειοψηφία. Να που έγκυται η λύση για τον backstop. Διότι εάν υπήρχε στενή σχέση, βαθιά όπως αυτή που περιέγραψε ο κύριος Μπαρνιέ, τότε το backstop θα υπάρχει. Αλλά δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί. Θα είναι θεωρητική διασφάλιση δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιείται καθημερινά. Οπότε και πάλι είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το είπε και ο κύριος Μπαρνιέτο και ο κύριος Γιούγκερ. Είναι στιγμή η πολιτική τάξη της Βρετανίας επιτέλους να πάει και σε αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα express, διότι εσείς θα πληρώσετε το τίμημα εάν δεν υπάρχει σαφήνεια. Η κυρία Σκοτ για τους ε, πρασίνους. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Westminster καταραίει. Έχουμε εσωτερικές αντιφάσεις λόγω του Brexit που ε, αναδύθηκαν χτες. Τελικά ήταν ένα σύνολο συνθημάτων. Ποτέ δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι σαν τη θέση προς διαπραγμάτευση. Ε, τώρα τελειώνει αυτή η ιστορία, ξεγυμνώνεται η υπόθεση και βλέπουμε όλες αυτές τις εφάνταστες ιδέες, αποτυχία. Και αυτό το χάος του Westminster σημαίνει ότι οι περισσότεροι Βρετανοί γνωρίζουν ότι το μέλλον της χώρας είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εδώ μπορούμε να συνεχίσουμε να, να, προς αυτό το όραμα που είναι το πιο αποτελεσμό για την ειρήνη, να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπερεθνικά ζητήματα όπως είναι το κλίματος, πρόκειται για την πλειοψηφία και οι νέοι ψηφοφόροι θέλουν να μας ψηφίσουν να βελτιώσουν την Ευρώπη μέσα σε κλίμα φιλίας, όλο ένα και περισσότεροι. Και τώρα έχουμε τους φουλευτές, απέρριψαν τον Οντίλ, άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις, πώς αυτό θα γίνει remain, πώς θα μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, να αποφασίσει ο λαός και η εχθρότητα αυτών που θέλουν τον Brexit. Τους βλέπουμε εδώ απέναντί μας. Ε, η εχθρότητα τους εναντί αυτών των δημοκρατικών αρχών σημαίνει ότι φοβούνται γιατί ξέρουν πως ξέρουμε και εμείς ότι η θέληση του λαού άλλαξε ε, άλλαξε το ρεύμα, όχι στο χάος του Brexit. Συνάδελφοι, αν μπορούσα, που δεν μπορώ, θα απαγόρευμα τη, τη λέξη βλαϊκή, σκουπίδια και δεν συμφωνώ μαζί σας που την είπατε κύριε. Λέει στον κύριο Φάρατζη, πρόεδρος. Σήμερα. Σας παρακαλώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα το, το, το ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε είναι να σεβαστούμε τον εκάστοτε ομιλητή. Έχουμε ένα σωρό ομιλητέ. Να και εδώ βλέπω προ τα δεξιά μου πάρα πολλοί, πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι παρεμβαίνουν. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι δυνατόν να το καταντήσουμε θέατρο εδώ στο Κοινοβούλιο. Ούτε είναι εδώ η Βουλή των Κοινοτήτων. Εδώ είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Danke. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φυσικά και σήμερα στην πολιτική μας ομάδα το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Τι θα κάνουμε σε σχέση με τη χτεσινή ψηφοφορία και την κατάσταση που έχει προκύψει και για μας ως πολιτική ομάδα τα πράγματα είναι σαφή. Εμείς στηρούμε, μένουμε στη συμφωνία για την αποχώρηση, που ήταν η μόνη εφικτή λύση. Δεν είναι το καλύτερο δυνατό που θα επιθυμούσαμε για να οικοδομήσουμε τις μελλοντικέ μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι αυτό που με μεγάλη ενέργεια, κόπο, απώλεια νεύρων πετύχαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο να εκπονήσουμε. Και κάποια στιγμή πιστεύω θα πρέπει κάποιος να αποφασίζει ε, αν αυτό που μπορεί να επιτύχει από κοινού με κάποιον άλλον, αν το τιμάει ή αν ο καθένας προσπαθεί από την πλευρά του να κερδίσει κάτι παραπάνω, να βγάλει κάτι και τελικά να ανατρέψει και να απειλήσει μαζικά ε, τα συμπεφωνημένα. Και θέλω να θυμίσω εδώ και ε, το λέω και εν ώψη των συναδέλφων ε, και υπόψη των συναδέλφων στο Ηνωμένο Βασίλειο, Συμβουλή των Κοινοτήτων. Πριν από δύο χρόνια περίπου, τι καταφέραμε, να έχουμε επιρροή στην εντολή που έλαβε ο κύριος Μπαρνιέ. Και στη συζήτηση αυτή μεταξύ άλλων καταφέραμε να καταδείξουμε πόσο σημαντικό είναι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός για να υπάρχει ε, πλήρως το θέμα ε, της ε, σταθεροποίησης της νευτικής διαδικασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά ήταν οι κόκκινε γραμμέ. Δεν ήταν τα δικά μα συμφέροντα, αλλά η σταθερότητα και η ειρήνη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αρχέ Γενάρη, στην πρώτη ψηφοφορία, είδα πολύ προσεκτικά τη συζήτηση και τη χθεσινή στη Βουλή των Κοινοτήτων και έχω την αίσθηση ότι δεν μα παίρνουν σοβαρά οι Βρετανοί μα συνάδελφοι. Και ορισμένοι δεν κατανοούν κάποιε διαδικασίε και συζητούν, λε και είναι οι μόνοι που θα ψηφίζουν για τι αλλαγέ. Αγαπητοί μου συνάδελφοι στο Λονδίνο, θα πρέπει να συζητήσετε και μαζί μας ε, για αυτά τα θέματα και να λάβετε υπόψη τη δική μας θέση. Δεν μπορεί να υποδίεστε ότι ισχύει η, η Βρετανική Αυτοκρατορία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε τη δική μας δημοκρατία. Μέχρι τώρα ήσασταν τμήμα της και πάντα φρόντιζα πάρα πολύ και εκτιμούσα πάρα πολύ ε, να ακούω αυτά που ήξερα από την Βρετανική διπλωματία και πραγματικά έχω φρίξει από αυτό το θέατρο που μας παίζουν. Είναι πολύ σημαντικό να επανέλθουμε, να επανέλθουμε στα βασικά και στα αυτά που θέλουμε τελικά να πετύχουμε και να μην περιχαρακωνόμαστε και κλεινόμαστε. Και η μόνη ελπίδα που έχω, το λέω, είναι στη συνεννόηση Corbyn May να υπάρξει κάποια μετακίνηση υπέρ των διαπραγματεύσεων με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μπορεί να λένε συχνά ότι είμαστε πρόθυμοι να έχουμε ε, συνεργασία. Αλλά αυτό που δεν θα κάνουμε, τουλάχιστον η δική μου πολιτική ομάδα και χαίρομαι που οι περισσότερες από τις άλλες ομάδες το βλέπουν αντίστοιχα και παρόμοια. Εμεί δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν να θυγούν τα εργασιακά δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά πρότυπα, η προστασία των ε, καταναλωτών, ούτε πιθαμή, πιθαμή δεν θα επιτρέψουμε η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής να μην γίνει σεβαστή ε, σε όλα τις τα τμήματα. Ούτε θα αφήσουμε κλειστά σύνορα στην Ιρλανδία. Ούτε να θεωρούνται πολίτες τρίτων κρατών ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και να υφίστανται διακρίσεις και να τους αφαιρούνται όλα τα δικαιώματα. Αυτό θέλω να το πω συνολικά στους συναδέλφους στη Βουλή των Κοινοτήτων. Τελειώνω. Χάρηκα όταν οι Βρετανοί συνάδελφοι πάλεψαν και απέκτησαν φωνή στη διαδικασία. Αλλά θα πρέπει να την ε, εκφράσουν και τη φωνή τους και δυνατά να μας πούν επιτέλους τι θέλουν. Κύριε Φαράζ, έχετε το λόγο. όλοι αυτοί, όλες οι ψηφοφορίες επηρεάστηκαν από το θυμό του κόσμου και είδαμε ότι δεν υπάρχει θέμα δεύτερη δημοσίευση. Τώρα έχουμε το άρθρο 50, δεν είναι πια ω επιλογή και ακούσαμε όλου του ομιλητέ να λένε ότι ανησυχούν και ότι έχει αυξηθεί το ρίσκο του no deal, έχετε δίκιο, μεγαλύτερο ρίσκο. Όχι όμω λόγω του, του ότι έγινε χθε το βράδυ, αλλά κύριοι, λόγω του των όσων εσεί είπατε τώρα, απόψε, ακόμα και όταν η Πρωθυπουργό συσπήρωσε μια πλειοψηφία, εντάξει, δέχομαι ότι έκανε ένα τερατώδες λάθος με τον προσυμπόραψη για το backstop και τέσσερα τα ξημερώματα έφυγε η Downing Street, πήγε ε, να, να σας βρει γιατί της βάλετε το τελεσίγραφο και επέγραψε κάτι που είναι ένα ναυάγιο. επέγραψε κάτι που καμία χώρα, εάν δεν έχει χάσει ένα πόλεμο, δεν θα υπέγραφε ποτέ. Ε, τώρα ε, συνειδητοποιούμε το λάθος και η Βουλή των Κοινοτήτων και όλη η χώρα τώρα αναζητούν μια συμφωνία. Ξέρετε όμως κάτι, πριν το δημοψήφισμα ουδής ήξερε ποια είναι, τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τίποτα, άγνωστη. Και τι είδαμε, ότι τώρα στην Βρετανία βλέπουν και εκτιμούν το ότι οι γρυφικάτες των ε, Βρυξελών ε, πείσανε, παρέπισαν, ε, ταπείνωσαν την Πρωθυπουργό και το λαό. δεν μας αρέσει αυτό και κάθε φορά που έρχεται και κάθεται για προμετεύσει, πως την είναι λογική και εσείς δεν υποχωρείτε ούτε ένα εκατοστό ε, να. Τώρα το Brexit είναι πιο κοντά. Και γιατί, λόγω της δικής σας γλώσσας, της στάσης σας, όχι μόνο της Κομισιόν, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι ε, του λαού, έναντι της χώρας μας. Και οπότε υπάρχει μεγάλο τιμός τώρα ε, έναντι των Βρυξελών. Και τι, τι θα έλεγε κάποιο. Ε, πρόκειται για φανατικού που δεν προτίθενται να δείξουν λογική. Κανένα συμβασμό δεν θέλουν. Και βεβαίω η Τερεζα συμβιβάστηκε ξανά και ξανά και ξανά. Ένα σωρό συμβασμοί παρασυμβιβάστηκε. Οπότε αρχίζουμε να λέμε το ότι ο κόσμο θα συνειδητοποιήσει ότι το no είναι καλύτερο από το backstop. Να το μεγάλο πρόβλημα για σας που θέλετε να επανεκλεγείτε σε λίγες εβδομάδες. Γιατί το no deal σημαίνει δεν θα υπάρχουν τα 39 δις. Πού θα βρείτε τα λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι τα 100 εκατομμύρια προσέκο που αγοράζουν κάθε μέρα από την Ιταλία θα ακριβίνουν. Και επίσης και όλα αυτά τα 750.000 γερμανικά αυτοκίνητα που αγοράζουμε. Άρα τι σενάριο ε, ετοιμάζουμε, γιατί ετοιμαζόμαστε να επικαλεστείτε το 24 ούτως ώστε όταν εμείς ε, φύγουμε τέλος του Μαρτίου να έχουμε δύο χρόνια χωρίς δασμούς, χωρίς ποσοστώσεις και περιορισμούς κανένας ε, είδους. Έχουμε προβλήματα, ή δυσκολίες με την Ιρλανδία, να έχουμε ξεμπλέψει με το Brexit και εσείς θα προστατευτείτε για δύο χρόνια. Α, οι ψηφοφόροι σας. Να, να ποιο είναι το επικοδομητικό βήμα που πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια ήταν μια μακρά και κοπιαστικότατη διαδικασία δυσκολιών, επανειλημμένων δυσκολιών που μας εμποδίζουν να εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως υπόθηκε και με το τρίκ, το βασικό αυτό τρίκ του backstop. Γι' αυτό απορρίφθη η συμφωνία και γι' αυτό επέστρεψε η κυρία Μέη να διαπραγματευτεί και πάλι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που όμω μα είπε δεν θέλει να διαπραγματευτεί. Υπάρχει ψηφοφορία από τη Βουλή των Κοινοτήτων για παράταση του άρθρου 50, όμω ξέρουμε ότι δεν γίνεται να συμβεί αυτό χωρί να συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα ζούμε όλοι για την 29η Μαρτίου. Θα τα καταφέρει το Βρετανικό πολιτικό ε, σύστημα να αποφύγει το δημοψήφισμα για δεύτερη φορά. Εάν δεν έχουμε συμφωνία στις 29 Μαρτίου και φύγουμε χωρίς πράξη αποχώρησης και εκτός κανόνου το άρθρο 50 δεν θα ισχύει πλέον, ούτε οι συνθήκες. Εάν η Βρετανική Βουλή δεν το αφήσει αυτό να συμβεί, είναι σαν να εξεγείρεται κατά του Βρετανικού λαού θα έχει βαθιές συνέπειες για οποιαδήποτε πίστη στη δημοκρατία που έχει απομείνει στον Ενωμένο Βασίλειο κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε ο κύριος Γούλφ. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τον Brexit. Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Βρετανική Δημοκρατία. Διότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια η κυβέρνησή μα έχει χάσει τον μπούσουλα. Αντί να διαπραγματεύεται αποτελεσματικά, ε, συμβιβάζεται και υποχωρεί ε, δείχνοντα αδυναμία. Θέλετε να μα παγιδεύσετε σε ένα μηχανισμό backstop που θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Όχι, δεν μπορείτε να μονοπολείτε το πολιτικό προσκήνιο του κόσμου. Θα πρέπει να δούμε τους συνεργάτες αυτού του σώματος και του Westminster που δεν μπορεί να αφήσει τους ε, υποστηρικτές του Ρημένα του Islington να πίνουν σαμπάνια στην υγεία της απουσίας συμφωνίας. Πέραν όλων αυτών και των αδυναμιών του νόμου, ο Βρετανικός λαός δεν θα σκύψει το κεφάλι. Δεν αισθανόμαστε φόβο, δεν ε, φοβόμαστε μια συμφωνία του ΠΟΕΡ, δεν φοβόμαστε ένα μέλλον ανεξαρτησία. Η Βρετανική κυβέρνηση επιτέλου κατάλαβε τι θέλει ο κόσμο και επιτέλου θα φροντίσει να απελευθερώσει το εμποριό μα. Καταλαβαίνει ότι η μάχη για αυτοδιάθεση, η ανεξαρτησία και η ελευθερία μα είναι τα βαθύτερα θεμέλια του έθνου μα. Θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε για να μπορέσουν αυτές οι πίστες μας να εκφραστούν ξανά ελεύθερα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το Brexit θα κάνουμε και θα ξαναγίνουμε ανεξάρτητη χώρα και πάλι. Ευχαριστούμε και τώρα για να ολοκληρωθεί η συζήτηση ο λόγος στην κυρία Τσιότ από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι σε περίπτωση που η κοινοβουλευτική διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο οδηγήσει σε κύρωση της συμφωνίας ε, ε, αποχώρησης, ελπίζουμε εντός προθεσμίας, θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα και θα αρχίσει η εφαρμογή της. Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να ε, παρακολουθείτε στενά έτσι ώστε να αποδώσει αποτελέσματα προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων και να συνεισφέρει στην εμπιστοσύνη που χρειάζεται για τις διαπραγματεύσεις των μελλοντικών μας σχέσεων οι οποίες ε, ε, μάλλον δύσκολες θα είναι. Ε, γι' αυτό προσβλέπουμε στη συνεργασία σας καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών αυτών τα επόμενα έτη. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Κλείνει εδώ αυτή η συζήτηση αγαπητοί συνάδελφοι.